Good evening uh, to all of... Καλησπέρα σε όλους σας για αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμών. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, θεωρούμε ότι η μερίσια διάταξη εγκρίνεται από όλους μας. Να προχωρήσω. Ωραία. Απόφαση των συντονιστών της 6ης Νοεμβρίου 2019 ε, θα τις βρείτε στους φακέλους της συνεδρίασης. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς αυτές, θεωρούνται και αυτές οι αποφάσεις συγκεκριμένε. Το ίδιο και για τα πρακτικά της συνεδρίασης της 6ης Νοεμβρίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται. Κυρία Χολμάγερ, η κυρία Χολμάγερ είναι καθοδόν. Όπου να είναι έρχεται για να μας ενημερώσει καλύτερα για το πώς πήγαν οι συζητήσεις της συνδιαλλαγής. Δεν θα το συζητήσουμε μέχρι να είναι εδώ. Οπότε θα έλεγα πρώτα να δούμε το διευθυντικό του προπολογισμού υπεριθμών 5, διότι ακόμα δεν έχει υποβληθεί σχέδιο έκθεσης, εφόσον το Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει ακόμα τη θέση του. Οπότε δεν γίνεται κι εμείς να εγκρίνουμε το διορθωτικό ή το διορθωτικό υπαριθμών 5 στην τρέχουσα Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Κύριε Χάουαρτ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχαμε ελπίσει ότι θα μπορέσουμε να το ψηφίσουμε αυτό το θέμα απόψε και ε, για μένα το θέμα ήταν αρκετά απλό, διότι πραγματικά το καθαρό ποσό του διορθωτικού είναι μόνο 1.900.300 ε, ευρώ. Οι αρχικές ενδείξεις που είχαμε ήταν ότι θα είναι ζήτημα διαδικαστικό, αλλά τελικά δεν πήγαν έτσι τα πράγματα. Το νωρίτερο που θα ψηφίσει για το θέμα αυτό το Συμβούλιο είναι την Πέμπτη. Και φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικοί αρκετοί λόγοι που ε, κάποια κάτι μέλη έχουν θέμα με την έκθεση αυτή, κάποιοι δεν έχουν μόνο τεχνικά ζητήματα, αλλά έχουν ε, λοιπά προβλήματα. Αυτό λοιπόν που προσπαθήσαμε να κάνουμε και να εισάγουμε δεν το καταφέραμε. Το διορθωτικό 5 είχε σκοπό να καλύψει κάποιες τεχνικές διευθετήσεις που χρειάζονταν ως προς την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ε, για το δημοσιονομικό έτος 2019. Δύο συμπεράσματα μπορούμε να διεξάγουμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση όπου το ένα θεσμικό όργανο λέει στο άλλο ε, στα πλαίσια της δημοσιονομικής διαδικασίας ότι εσύ πρέπει να συμφωνήσεις με μια συγκεκριμένη πρόταση θες δεν θες. Το ε, κοινοβούλιο δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ούτε και το συμβούλιο, διότι προφανώ η δημοκρατική ε, εξέταση του προπολογισμού δεν θα είχε κανένα νόημα. Και επίση είναι ατυχέ που έχουμε βρεθεί στη θέση και ίσω γι' αυτό θα πρέπει να περιοριστούμε απολύτω τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Brexit, στην Συμφωνία Κυρίων. Τη Συμφωνία Κυρίων μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ε, κάτι που προέβλεπε ότι δεν θα ασχολούμαστε ένα με τον προπολογισμό του άλλου ή δεν θα τον ε, εξετάζουμε ξενυχιστικά. Πράγμα που θα διέπει και το διορθωτικό υπαριθμών 5. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή θα πρέπει να εργαστεί σκληρά για να βεβαιωθεί ότι θα βρεθεί μια θέση ισορροπία και για τέτοιου είδου περιπτώσει. Κύριε Πρόεδρε, ίσω ήταν χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα ε, πει την άποψή τη για το πώ βλέπει τα πράγματα σε σχέση με το διορθωτικό 5. Κάποιος από τους σκιώδεις εισηγητές θέλει να προσθέσει κάτι. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ρέιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον κύριο Χάουαρτ που εισήγαγε το θέμα. Όντως, το θέμα του διορθωτικού του προπολογισμού επαριθμών 5 ε, υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα το διορθωτικό υπήρξαν κάποια σχόλια και το Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα επανεξετάσει το διορθωτικό την Πέμπτη. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί παρά να προσπιστεί την πρόταση την οποία επέβαλε και δεν μπορώ να προδικάσω τι θα πει το Συμβούλιο την Πέμπτη. Οπότε είδομεν. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι το θέμα θα έπρεπε να είναι πραγματικά απλό, αυτόματο. Οι επιπτώσεις του Brexit για τα θεσμικά όργανα και λόγω της αναβολής του Brexit, οι επιπτώσεις της ε, μισθολογικές προσαρμογές στα θεσμικά όργανα είναι το νέο στοιχείο του σκέλους για, τα, για τους μισθούς στο διευθυντικό του προπολογισμό. Καταλαβαίνω καλά κύριε Ρέιλ, είναι τεχνική η λόγη της καθυστέρησης. Θα το δούμε την Πέμπτη. Είναι αρκετά πιθανό, άρα το Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφασίσει ότι θέλει να συντομεύσει την περίπτωση εξέταση των 8 εβδομάδων από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα και αυτό είναι ένα τεχνικό λόγο. Κατά τα άλλα, δεν είμαι απολύτω βέβαιο. Ωραία. Εάν δεν είστε βέβαιο, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι κι εμεί. Κύριε Χάουαρτ, θέλετε να μα διαφωτίσετε περαιτέρω για τα επόμενα βήματα. Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη. Ωραία. Ευχαριστώ. Sorry. Με συγχωρείτε, κυρία Χολμάγερ δεν έχει φτάσει ακόμη, οπότε να προχωρήσουμε με την εμερήσια διαταξή μας και θα έλεγα να περάσουμε στη συζήτηση των, ε, της έκβασης της συνδιαλλαγής. Νομίζω ότι όλοι όσοι συμμετείχαν Αξίζουν συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα που πετύχαμε. για την αύξηση στα 850.000 εκατομμύρια, των οποίων μεγάλο 850 εκατομμύρια, εκ των οποίων μεγάλο μέρος στην έρευνα και την ανάπτυξη και τα σχετικά ζητήματα. Νομίζω ότι παραμείναμε συσπηρωμένοι ως ομάδα, εισηγητές και σκιώδης εισηγητές. Εργαστήκαμε σκληρά και ήταν αρκετά παράξενο που μετά από συζητήσεις, για να το πω έτσι και αρκετά έντονες κάποιες φορές με το Συμβούλιο, διαβάσαμε μετά το δημοσίευμα τύπου του Συμβουλίου, που είδαμε να χρησιμοποιεί κάποια επιχειρήματα το Συμβούλιο για να πει ότι η συνδιαλλαγή ήταν επιτυχημένη. Ευχάριστο να το βλέπει κανείς από αυτή τη σκοπιά. Κυρία Γκοροντιαδεχαμπάλ, θέλετε να πείτε κάτι για τα αποτελέσματα και πώς τα πετύχαμε και οποιοδήποτε από τους υπόλοιπους συνεισηγητές. Κυρία Γκοροντιαδεχαμπάλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον αρκετοί, είμαστε στην ε, συνδιαλλαγή. Τελικά νομίζω ότι καταλήξαμε σε καλό αποτέλεσμα και ξεχνάμε τις απογοητεύσεις κάποιων. Αυτό είναι σύνηθες. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη ότι είχαμε πολύ διαφορετικές εξ αρχής θέσεως με το Συμβούλιο, με μαξιμαλιστικές εκ μέρους μας και μινιμαλιστικές θέσεις εκ μέρους Συμβουλίου, βρήκαμε την ε, μέση λύση, τη χρυσή τομή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι όντως το Συμβούλιο κατανόησε ότι δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια περικοπές στον ε, προϋπολογισμό μας και μπορέσαμε και να ενισχύσουμε για τις προτεραιότητές μας ίσως το πιο σημαντικό σημείο εκτός από τους αριθμούς που όντως μπορούμε να δούμε θετικά είναι πως αντικατοπτρίστηκε όλο αυτό το εγχείρημά μας στον τύπο, με θετικό τρόπο. Και βεβαίως στον ε, ισπανικό τύπο αυτό είναι προφανές και τονίζεται και ίσως και σε άλλες χώρες ότι ένα στα πέντε ευρώ αφιερώνεται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο θέσαμε τις προτεραιότητες για το 2020, αλλά και για όλο το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε το όλο θέμα. Ε, εγώ ήμουνα για ενδέκατη φορά και πρέπει να πω ότι ήταν η καλύτερη και χάρη στο Κοινοβούλιο και στη Γραμματεία και σε εσά που εργαστήκατε πάρα πολύ, αλλά και επειδή έκανε πολύ σοβαρή δουλειά και η Φινλανδική Προεδρία τη στιγμή που έπρεπε να οργανώσει διαπραγμάτευση, πολύ οργανωμένα τι ώρα, τι ώρα θα κάνουμε τη συνεδρίαση, πότε θα συναντήσουμε επιμέρους τις διάφορες ομάδες, πότε θα φτάσει η Επιτροπή να μας παρουσιάσει στους ε, Συμβούλιο και σε εμά ε, τις θέσεις της, μας βοήθησε, έγινε με τέτοιο τρόπο που μας βοήθησε να μην έχουμε παρανοήσεις και προβλήματα και μπορέσαμε με αυτό το ρυθμό, τον πάρα πολύ καλά οργανωμένο, να τις ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις, διότι διευκολύνθηκε πάρα πολύ όλη η διαδικασία χάρη στην οργάνωση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τη Γραμματεία, τη Μόνικα που δεν είναι εδώ, η οποία επιτέλεσε εξαιρετική εργασία, διότι όπως και εσείς και εγώ κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρουμε είμαστε παρόντες σε όλες τις συνεδριάσεις και ξέρουμε ότι υπερασπίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Μόνικα τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτοιμοι λοιπόν για να μπορέσουμε να εργαστούμε και για του χρόνου για τον προπολογισμό. Τέλο πάντων, εγώ λέω το κομμάτι το οποίο με αφορά. Πρώτον, πρέπει να πω ότι αποφύγαμε οποιοδήποτε πρόβλημα με τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν ο στόχος μας. Δεύτερος, πρέπει να πω ότι ξεκινήσαμε, ίσως όχι με το δεξί, αλλά κατά τη διάρκεια της συνδιαλεγής είδαμε ότι πραγματικά μπορέσαμε και κάναμε καλή διαπραγμάτευση. Τώρα, με άλλα τμήματα, όπως πάντα, είναι δύσκολο να τα πετύχουμε όλα. Όχι ότι δεν επέμεινα, αλλά ξέρουμε ότι αν ανοίξουμε διαπραγματεύσεις για άλλα τμήματα, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε την πόρτα στο Συμβούλιο που θα, αρχίσει, θα άρχιζε ενδεχομένω να κάνει χιλιάδες ερωτήσεις για το πώς διοικούνται οι μεν και οι δε. Μπες περιπτώσει κάποια τμήματα λοιπόν που δεν ήταν της δικής μας της αρμοδιότητας τα αφήσαμε και έτσι αποφύγαμε περικοπές που ήθελε να κάνει καταρχά το Συμβούλιο. Πρέπει λοιπόν να πω ότι ίσω δεν καταλήξαμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στην ε, καλύτερη δυνατή διαπραγμάτευση, αλλά μπορέσαμε να διαπραγματευτούμε ένα αξιοπρεπές προϋπολογισμό και για τα άλλα θεσμικά όργανα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίω. Σας ευχαριστώ. Κύριε Φερνάντες. Θα ήθελα να συγχαρώ την Μόνικα και την κυρία Ρζαμπαχλά, καθώς και όλους τους ε, σκιώδεις που είπαν ναι στην ε, συμφωνία και να πω επίσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, στη γραμματεία, στους συμβούλους, σε όλους όσοι συμμετείχαν. Είχαμε εξαιρετικό αποτέλεσμα που είναι αποτέλεσμα και της ενότητας που βλέπουμε ότι υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε ενωμένοι και επιτύχαμε. Πρόκειται λοιπόν για πολύ καλό παράδειγμα και για άλλους φακέλους, κυρίως για το πολιωτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βεβαίως και η Προεδρία πρέπει να πω και το Συμβούλιο πέδειξαν ότι υιοθέτησαν μια πολύ λογική στάση. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτά τα οποία λέξαμε για το πολιετές στον τύπο θα επαληθευτούν. Δηλαδή αν προς, μας προσεγγίσουν θα μπορέσουν να κάνουν και ε, διά, να πείσουν και τον τύπο ότι έχουν θετική άποψη. Τα θέματα της, ε, της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας, της απασχόλησης, ε, της ε, έρευνας για την καταπολέμηση του καρκίνου. Όλα αυτά είναι θέματα προτεραιότητας και επιμένω όντως αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένα από τους καλύτερους του Κοινοβουλίου. Πρέπει να πω ότι και εγώ είμαι 11 χρόνια Ευρωβουλευτής και επαναλαμβάνω και πάλι τις ευχαριστίες μου σε όλους όσους μετήχαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μπορούμε να το επαναλάβουμε αυτό. Βεβαίως, πρέπει να πω ότι ούτε κάθε πολιτική ομάδα, ούτε καθένας από μας είδε όλες του οι προτεραιότητες να ικανοποιούνται, αλλά τουλάχιστον επιτύχαμε μια εξαιρετική ισορροπία και οι πολίτες μπορούν να συνεχίζουν να υπολογίζουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών να θεωρούνται δεδομένες τώρα μετά τη θεωρία μας μένει να τις θέσουμε σε, στην πράξη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω αυτά που είπε και η Αντέρ και ο Ξεμανουέλ λένε ότι είναι δέκατη, δεκατη φορά συνάδελφοι, ντρέπομαι. Εμένα ήταν η πρώτη μου φορά, αλλά πρέπει να πω ότι όλοι μαζί συνεργαστήκαμε ε, και είχαμε καλά αποτελέσματα. Είχαμε μεγάλες φιλοδοξίες και πίστευα ότι θα φανεί ότι είμαστε γελοί. Στο τέλος όμως αυτό το αποφύγαμε διότι είδαμε και τις πέντε πολιτικές ομάδες να υπάρχει ενότητα. Είδαμε, όπως είπε και ο Χωσέ Μανουέλ, ότι όλοι μαζί υπερασπιστήκαμε την ε, καταπολέμηση ανεργία των νέων, την απασχόληση για τους νέους. Βεβαίως θα θέλαμε περισσότερα πράγματα, βεβαίως είναι ανεπαρκές αυτό που έγινε για να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των ε, πολιτών και των κοινωνιών μας για την κλιματική αλλαγή, αλλά πρέπει να πω ότι κάτι κάναμε. Πολλοί από εμά είναι καινούργοι και αυτή η δουλειά, η συλλογική που επιτελέστηκε μας δίνει όρεξη να συνεχίσουμε. Η επόμενη μάχη, αλλά συμφωνούμε, είναι να μπορέσουμε να βρούμε νέους πόρους. Διότι όλοι θέλουν περισσότερη Ευρώπη, αλλά όπως θα θυμάστε και η κυρία Θάτσερ έλεγε όχι με τα λεφτά μου, όχι με τα λεφτά μου. Πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες λοιπόν για κοινωνικά θέματα, για έρευνα θα πρέπει να έχουμε ε, περισσότερους πόρους. Εγώ ήμουν νέος όταν έλεγε ο Ζακ Ντολόρ πριν από 20 χρόνια ότι χρειαζόμαστε δύο σπόρους δικούς μας, όντως ισχύει αυτό πάντα. Ευχαριστούμε τους πάντες, τους συναδέλφους, τη γραμματεία και τους εμπειρογνώμενους δικούς μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο? Ευχαριστώ πολύ. Ήδη έχουν αναφερθεί τα περισσότερα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εισηγητές και τη Μόνικα Χολμάιερ και την ε, κυρία Γκαρδία Θάμπαλ για την εξαιρετική δουλειά τους, αλλά και εσά, ε, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως ε, καλώς δείξαμε την δύναμή μας και την ε, ξεκάθαρη θέση μας ως ε, Κοινοβούλιο. Έχουμε συζητήσει για το ότι η θέση μας πρέπει να είναι ισχυρή, γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ήταν καλό που είχαμε μια ισχυρή εντολή έτσι ώστε να μπορέσετε να διαπραγματευτείτε εκ μέρους μας. τα μέσα ενημέρωσης ήταν θετικά στη Γερμανία και είδαμε ότι και άλλα κράτη-μέλη ήθελαν να κάνουν περικοπές, όμως δεν είχαν καλά επιχειρήματα. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη θέση μας δημόσια, να έχουμε μια καλή ανταλλαγή απόψεων, μια ισχυρή διαβούλευση έτσι ώστε να διαπραγματευτούμε το προεπιλεσμό του 2020. Όμως ε, για μας τους πράσινους ε, πρέπει να συνεχίσει η δουλειά, πρέπει να πάμε ακόμα παραπέρα, να διαπραγματευτούμε ενωμένοι για τις κοινέ μας θέσεις. Και χρειάζονται περισσότερα κονδύλια για το κλίμα όταν θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέλουμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, αλλά γι' αυτό πρέπει να δείξουμε και αποτελέσματα. Πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε πως ε, αυτό είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά νομίζω πως είναι στο χέρι μας να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, τότε νομίζω πως μπορούμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Να αναφέρω επίσης ότι η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τον προϋπολογισμό θα λάβει χώρα, αν δεν κάνω λάθος, την Τετάρτη. υπομονούμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Ας ελέγξουμε αν λειτουργούν τα συστήματα. Νομίζω πως όλα πρέπει να είναι εντάξει. I the vote open. Please vote that we can... Ας ψηφίσουμε λοιπόν για να δούμε αν όλα λειτουργούν. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Κύριε Πρόεδρε, ξέχασα την κάρτα μου στο μηχάνημα της αίθουσας Ολομέλειας, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να το λάβω την υπόψη. Okay. We count you on top as we proceed. Ωραία, θα δούμε στην πορεία. Ξεκινάμε με την πρόταση απόφασης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του ε, μηχανισμού του Ταμείου Αλληλεγγύης για την πληρωμή προκαταβολών στον Γενικό Προϋπολογισμό για το 2020. Άρχεται η ψηφοφορία. Declare the vote closed. Πέρας. Συν μία ψήφος για τον κύριο Χόουαρθ. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Περνάμε στην πρόταση κινητοποίησης του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των ισρών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας. Ξεκινάμε με τις τροπολογίες. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 θα εξεταστούν μαζί με ανάταση των χεριών. Ποιο είναι υπέρ, ποιο είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση για την πρόταση. Άρχεται. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα. Έχουμε και εδώ τροπολογίες. Ξεκινάμε με την τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δεν υπάρχουν αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το τελικό κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας Αλληλευτικής Σύμπραξης. Θα εξετάσουμε και τον ε, εφιστάμενο φάκελο και τον επόμενο για την ε, Γουινέα Μπισάου και για τη δημοκρατία του Σάτομε και Πρίνσιπε. Έχουν παρουσιαστεί και συζητηθεί μαζί στις 26 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Αλία. Να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για διαδικασία συνένεσης, άρα ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία για την πρώτη συμφωνία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στο δεύτερο πρωτόκολλο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο. Νομοθετική πρόταση για τους, τις μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Δοτική Ανάπτυξης. Η Επιτροπή ε, Γεωργίας είναι η καθήλυνα αρμόδια για το σύνολο. Τη δέσμη μέτρων αποτελείται από δύο προτάσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία, έτσι ώστε να δοθεί παράταση και να συνεχίσει να ισχύει για το 2020 και 2021 χωρίς νομική ασάφεια. Αυτό είναι αναγκαίο διότι η διαδικασία ναι, διαπραγματεύσεων, όπως γνωρίζετε, εξελίσσεται πάρα πολύ αργά. Δεν υπάρχει πρόοδος στους τρεις κανονισμούς που θα αποτελέσουν το ε, κομμάτι για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι συντονιστές αποφάσισαν την ε, περασμένη εβδομάδα ότι θα γνωμοδοτήσουμε για τους δύο φακέλους και μια που η Επιτροπή Γεωργίας πρέπει να ψηφίσει ήδη στις αρχές Δεκεμβρίου με την επισπεσμένη διαδικασία, οι γνωμοδοτήσεις αυτές θα δοθούν με τη μορφή επιστολής από τον Πρόεδρο. Έχουν αποσταλεί την περασμένη εβδομάδα σχέδια στις πολιτικές ομάδες, έχουν λάβει την έγκριση των συντονιστών, διότι υπάρχει ένας ε, στόχος ε, να έχουμε κοινή προσέγγιση. Δεν χρειάζεται φυσικά να βλάψουμε λόγω της βιασύνης μας το τελικό αποτέλεσμα και να ζημιωθούν τελικοί δικαιούχοι. Ψηφίζουμε τώρα στις, για τις δύο επιστολές. Για την πρώτη επιστολή, η οποία σας διαναμήθηκε σήμερα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνατε. Ψηφίζουμε την γνωμοδότηση για τις μεταβατικές διατάξεις, επίσης με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο, μεταφορές, τμήμα 3, κύριε Χόουαρθ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μόνο μία μεταφορά εξετάζουμε σήμερα στον Γενικό Προϋπολογισμό. Αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον, μία διαφορά που έχει προκύψει από τις διαφορές στο άπαχο γάλα. Έπειτα κάποιες μειώσεις για τα κονδύλια που δεν έχουν δαπανηθεί. 951.200 ευρώ. Το ποσό αυτό προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για την γραμμή του προϋπολογισμού όπου η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την ε, προσφορά. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, σε γενικές γραμμές για το πρασίνισμα της γεωργίας. Αυτό θα μας επιτρέψει και να εκπληρώσουμε τους στόχους μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 67 463 67.463.000. Η Κομισιόν θέλει να σχολιάσει, όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο μεταφορέ το 2019, υπόλοιπα τμήματα. Κύριε Φερνάντε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα τα πω πορτογαλικά. Έχω τέσσερις μεταφορές από τον προπολογισμό για τα υπόλοιπα τμήματα. 30.000 ευρώ για, τη, για, την, για τους υπολογιστές και τις τηλεπικοινωνίες, και 200.000 ευρώ επίσης γι' αυτό μετά 50.000 ευρώ για τις ψηφιακές και παραδοσιακές δημοσιεύσεις. Σκοπός της μεταφοράς αυτής είναι η τεχνολογική υποστήριξη προς τους ευρωβουλευτές ε, ως συνέπεια των εκλογών του 2019 και έχει να κάνει και με την υποβολή μάλλον με τη νέα εφαρμογή, τη νέα, το νέο εφαρμογή στο ίντερνετ ή petition και την ε, συντήρηση του Κοινοβουλίου. Επίσης, για τα στοιχεία 2140 και 3200 ε, είχαμε εξοικονομήσεις, γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ της συγκεκριμένης μεταφοράς. Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω πορτογαλικά. Ε, πρότεινα να ψηφίσουμε υπέρ της μεταφοράς αυτής. Τώρα για την επόμενη, για τις δύο επόμενες. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε υπέρ, αλλά δεν ξέρω αν έχει κάτι να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία, συνεχίζω. Ε, για την ε, Μεταφορά ε, C17. Εδώ θέλαμε να υποστηρίξουμε τις δαπάνες των τομέα των οπτικοακουστικών 1.400.000. Ο στόχος της μεταφοράς είναι να δώσει χρηματοδότηση για την τρίτη και τελευταία φάση της ανανέωσης του επικοκουστικού εξοπλισμού στο Στρασβούργο. Η μεταφορά αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί χάρη στις εξοικονομήσεις που έγιναν στο σημείο του 3000, ε, έξοδα για τις ε, αποστολές και τα ε, υπηρεσιακά ταξίδια μεταξύ των τριών εδρών. για αυτήν την ε, μεταφορά που έχει αξία 1.400.000 ευρώ ήθελα κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Θα χρειαζόντουσαν περισσότερες πληροφορίες για να μπορέσουμε να την εγκρίνουμε. 1.400.000 ε, ευρώ. Ο κύριος Καρμπάχο είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Η ε, επιπλέον Η μεταφορά αυτή έχει να κάνει με μια δουλειά που έγινε επί τέσσερα έτη για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον εξοπλισμό των οπτικοακουστικών του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Έχουμε φτάσει σε αυτή την τελική φάση, όπω είπατε, γιατί πρέπει να υποστηρίξουμε τι υπηρεσίε που προσφέρονται προ του βουλευτέ. Είναι μια δουλειά ε, υποδομή που δεν τη βλέπουμε, δεν είναι τόσο ορατή, με σερβερ, με άλλα τεχνολογικά στοιχεία, για να μπορέσουμε μέχρι το 2020 να έχουμε όλα τα στοιχεία στι εγκαταστάσει που χρειαζόμαστε, όπω το Boxbox και άλλα πολλά που ξέρετε από τι Βρυξέλλε, τα θέλουμε και στο Στρασβούργο. Ε, είναι όλα αυτά εγκαταστάσεις που έχουν να κάνουν με το ημικύκλιο, με την αίθουσα της Ολομέλειας, το πώς ε, εργάζονται οι εκπρόσωποι του τύπου. Και επειδή θέλουμε όλες αυτές οι υποδομές να είναι έτοιμες το 2020, θέλουμε να μπορούμε να προσφέρουμε τι ανάλογε υπηρεσίε στου ευρωβουλευτέ, τι άμεσε και έμεσε υπηρεσίε και έχει να κάνει και με τη συνεργασία μα με του εκπροσώπου του τύπου. Μιλάμε για τον χώρο των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και ακριβώ η φετινή ε, χρονιά απέδειξε ότι είναι ο καλύτερο τόπο για να παράσχουμε στου βουλευτέ αυτέ τι επιπλέον υπηρεσίε που χρειάζονται. Με πιστώσει που δεν καλύπτονται από τον τρέχοντα προπολογισμό, μιλάμε για κονδύλια που είχαν να κάνουν πιο πολύ με συντήρηση, αλλά όχι με νέε εγκαταστάσει. Ωραία. Με τις εξηγήσει αυτές λοιπόν νομίζω μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ. Τώρα για την μεταφορά C18 θα συνεχίσω πάλι στα πορτογαλικά. Η μεταφορά αυτή σκοπό έχει να ενισχύσει το στοιχείο 2102, υπολογιστές και τηλεπικοινωνίες και γενική υποστήριξη των χρηστών με 223.500.000 ευρώ και στο στοιχείο 2104 υπολογιστές και τηλεπικοινωνίες επενδύσεις στις υποδομές 4.661.500 ευρώ. Σκοπός της μεταφοράς αυτής είναι να προσφέρει ε, χρηματοδότηση και να επιτρέψει να γίνουν επενδύσεις ε, για τους υπολογιστές του data, του κέντρου δεδομένων του Κοινοβουλίου και να αυξηθεί το επίπεδο τεχνολογικής υποστήριξης προς τους βουλευτές μετά τις εκλογές του 2019. Ήθελα και εδώ κάποιες περισσότερες πληροφορίες για, το, για τη συγκεκριμένη μεταφορά αυτή στον προπολογισμό. Μάλιστα, ο Γενικός Διευθυντής της TGI Tech έρχεται, ψάχνει που να καθίσει, καθίστε κάπου, Make yourself... βολευτείτε και πείτε μας. Να πω ότι αναφερόμουν στο C18 και στη μεταφορά των 4.661.500 ευρώ. Ήθελα εδώ επιπλέον πληροφορίες. Υπολογιστές, τηλεπικοινωνίες και επενδύσεις στις υποδομές. Ήθελα κάποιες εξηγήσει για, το, για τη μεταφορά αυτή. Κύριε Πατρότσι, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, έρχομαι από την ε, συνεδρία του Προεδρείου. Να με λοιπόν. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας κύριε Φερνάντες σε ό,τι αφορά το έμβασμα αυτό, τη μεταφορά C18. Είναι τρία τα σκέλη. Το ένα ε, αφορά ένα ποσό 250.000 περίπου ευρώ για την υποστήριξη των ευρωβουλευτών. Μιλάμε για μια διαρθρωτική ε, υποστήριξη, μια υπηρεσία που προσφέρει υπηρεσία, που συνοδεύει τους βουλευτές στη δουλειά τους, δημιουργήθηκε φέτος και σκοπό έχει να προσφέρει περισσότερα στους βουλευτές. Ε, υπηρεσίες εγκύτητας και αντιδραστικότητας, για να το πω έτσι. Θέλουμε δηλαδή ουσιαστικά να φουγκραζόμαστε τις ανάγκες των βουλευτών, να κατανοούμε καλύτερα τη δουλειά τους και να μπορούμε ε, στοχευμένα να υποστηρίξουμε όσα κάνουν. Ε, μιλάμε για ένα πρόγραμμα κατάρτισης κιόλας εδώ, ε, στα του, πρόεδρου της υπηρεσίας, και αυτό αφορούν αυτό το ποσό. Τώρα έχουμε, λέμε για δύο μεγαλύτερα ποσά. Το ένα είναι των 2 εκατομμυρίων επενδύσεις που θέλουμε να κάνουμε ε, στο κέντρο δεδομένων, το data center, για να γίνουν τα συστήματα λίγο πιο εύρωστα. Να υπάρχει μια συνέχεια στην προσφορά υπηρεσιών και να είναι διαρκώς διαθέσιμα. Να υπάρχουν πληροφορι... υπηρεσίες πληροφορικής και IT 24 ώρες, 24 ώρα, 7 μέρες τη βδομάδα. Εδώ θέλουμε να ενισχύσουμε ακριβώς αυτή τη διάσταση για να γίνουν τα συστήματα πιο αξιόπιστα και να υπάρχει η διάρκεια στην προσφορά των υπηρεσιών χωρίς διακοπές. Υπάρχει κι άλλο ένα στοιχείο για τις ε, αγορές που θέλουμε να κάνουμε και να αξιοποιήσουμε το cloud, το υπολογιστικό νέφος. Απόφαση που ελήφθη φέτος από το Προεδρείο, απόφαση που θα μας επιτρέψει να απλώσουμε τα πλοκάμια μας ως data center προς το cloud, ε, προς το υπολογιστικό νέφος, δηλαδή να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας και την ε, ελαστικότητα που διαθέτουμε για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε υποδομές ε, για τους για τους παρόχους και για τους ευρωβουλευτές. Ε, ε, για τους βουλευτές επίσης υπάρχει και το θέμα της ε, κινητικότητας, δηλαδή θέλουμε να τους προσφέρουμε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους για να μην έχουμε κενό εκεί. Αυτό για τα 2 εκατομμύρια και μετά έχουμε τα 2,5 εκατομμύρια που ζητούμε. Αυτό σκοπό έχει να αντιμετωπίσει την παλαιότητα των συστημάτων. Δηλαδή έχουμε εγκαταστήσει κάποιου υπολογιστέ που κάποια στιγμή ξεπερνιούνται από τις εξελίξεις. Ε, πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα προγραμματισμό εγκαίρος για την αγορά νέων, αλλά το ποσό αυτό το ζητούμε διότι τη χρονιά νη 2, το 2017 ήδη είχαμε ετοιμάσει τον προπολογισμό το 2019 και τότε έπρεπε να περιορίσουμε λίγο την ζήτηση και να παραμείνουμε σε, σε στα όρια της εύλογης, ζήτησης. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συστηματικά στο πλαίσιο των δεσμικών οργάνων. Μιλάμε λοιπόν για ένα κονδύλι το οποίο πρέπει να διατεθεί τώρα και να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες αγορές για να αντικαταστήσουμε τα μηχανήματα που είναι πλέον ε, απερχιωμένα. Έχουν ξεπεραστεί. Ευχαριστούμε κύριε Φερνάντες. Ωραία λοιπόν και εδώ ευνοϊκή ψήφος. Τώρα το επόμενο. Η επόμενη μεταφορά στον προπολογισμό είναι τη Επιτροπής των Περιφερειών, το ΙΝΦ4. 2019 ε, με σκοπό ε, να ασχοληθεί με την ανανέωση ε, των τεχνολογικών εγκαταστάσεων Λίμα 2007 208.000 ευρώ και το 2100 IT ε, λογισμικά και υπολογιστές, 102.000 ευρώ. Αυτά είναι απαραίτητα για την ανανέωση των τεχνολογικών εγκαταστάσεων για τους συναδέλφους του Επιτροπής των Περιφερειών με χρηματοδότηση που δεν ήταν ε, αρχικά διαθέσιμη στον προπολογισμό της Επιτροπής. Η μεταφορά αυτή χρηματοδοτεί επιπλέον προγράμματα και προβλέπεται από τις δεσμεύσεις του INF3 2019. Τα επιπλέον αυτά προγράμματα ε, καλύπτονται από κοινού από τον Διεύθυνση για την ε, για τη λογιστική, για την επιμελητία του, της Επιτροπής των Περιφερειών και της ε, Της, της ΕΟΚΕ. η, μεταφορά που μας μένει είναι η VAB 18T19, η οποία σκοπό έχει να υποστηρίξει το ε, 2100 με 150.000 ευρώ για την αγορά ε, και την συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού και το στοιχείο 2008, μελέτες και τεχνική υποστήριξη σε σχέση με σχέδια οικοδόμησης, 25.000 ευρώ, καθώς και το στοιχείο 2026, ασφάλεια και παρακολούθηση των κτηρίων και με 100.000 ευρώ και το 2022 για υπηρεσίες καθαριότητας και συντήρησης 25.000 ευρώ. Η μεταφορά αυτή σκοπό έχει να υποστηρίξει την εικονική υπηρεσία μεταξύ δύο κέντρων δεδομένων που ε, αφορούν το ελεγκτικό, το ελεγκτικό συνέδριο και πρέπει να εγκριθούν για να μην παρεμποδιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Και εδώ ευνοϊκή αποτίμηση και αυτά λίγο πολύ ήταν τα συναρπαστικά του θέματος των μεταφορών στον προπολογισμό. Ευχαριστούμε. Κύριε Στεφανούτα, με συγχωρείτε, δεν θα έπαιρνα το λόγο για το σημείο αυτό, γιατί συνήθω οι μεταφορές ε, πηγαίνουν ρολόι, αλλά ήθελα να πω κάτι για το προηγούμενο σημείο, για, αφού κάναμε εξοικονομήσεις. Επειδή οι βουλευτές δεν προσέλαβαν αυτές τις αρκετούς βοηθούς, Ήθελα να ρωτήσω τον διευθυντή που είναι εδώ μαζί μα, γιατί δεν επενδύουμε αυτά τα χρήματα στο σχέλο τη κυβερνοασφάλεια των υποδομών, των υποδομών που ήδη χρησιμοποιούμε σε αυτό το σώμα. Διότι υπήρξαν ε, ειδήσει ότι παρατηρήθηκαν παραβιάσει στο σύστημα κυβερνοασφάλεια, ότι διέρευσαν πληροφορίε και στη συζήτηση που θα γίνει αυτή την εβδομάδα στην Ολομέλεια για τις ε, παρεμβολές από τρίτα κράτη στο δημοκρατικό μας ε, οικοδόμημα, φαίνεται να υπάρχουν ε, πολλά τέτοια θέματα. Θέλω λοιπόν το θέσω και αυτό ε, υπόψη σας, για τις μεταφορές στον προπολογισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τις μεταφορές που μας παρουσίασε ο κύριος Φερνάντε, θεωρούμε ότι μπορούν να εγκριθούν. Εντάξει, υπάρχουν αντιρρήσεις. Ευχαριστώ. Building policy. Ως προς την πολιτική των κτηρίων δεν υπάρχουν θέματα προς ψήφιση. Νομίζω ε, συμφωνείτε με αυτό όλοι. Κλείνουμε εδώ το σημείο για τις προφορίες και έχουμε ένα τελευταίο σημείο, το πρωτόκολλο για την υλοποίηση της αλληλευτικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Δημοκρατίας του Πράσινου Ακροτηρίου. Κυρία Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία μεταξύ του στις του Πράσινου Αγροτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε στι το 2007. Το πρώτο πρωτόκολλο τέθηκε σε εφαρμογή το Δεκέμβρη του 2014 και το Δεκέμβρη του 2018 έλξε στο μεταξύ διάστημα έκανε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση ε, της χώρας αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συνάψει νέο πρωτόκολλο συμφωνίας με στόχο να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην δημοκρατία του Πράσινου Ακροτηρίου να συνεργαστούν περισσότερα ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν με βιώσιμο τρόπο τους αλληλευτικούς πόρους του, του πράσινου ακροτηρίου να επιτρέψουν στη χώρα αυτή να αναπτύξει περισσότερο την ε, οικονομία της. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της πολιτικής αλληλείας, αυτό το νέο πρωτόκολλο δίνει δυνατότητες αλληλείας στον αλληλευτικό στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα χωρικά ύδατα της δημοκρατίας αυτής. Σύμφωνα με τις ε, συστάσεις της ε, ε, διεθνούς οργάνωσης για την ε, διατήρηση και τη διάση των ηλεκτρικών πόρων. Αυτό είναι μέρος της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα κράτη ΑΚΕ. Λαμβάνουμε υπόψη κυρίως τους αντικειμενικούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει την διασφάλιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, στις εξής κατηγορίες προβλέπεται ε, συμφωνία. 28 ε, αλευτικά σκάφη τόνου, 17 ε, τράτες και λοιπά αλευτικά σκάφη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέχει 750.000 ευρώ ώστε να μπορέσουν να αλλιεύονται 8.000 ε, τόνοι αλλιευμάτων κατά τη διάρκεια της ισχύω του πρωτοκόλλου και δεύτερον υποστήριξη στην ε, ε ανάπτυξη της αλλιευτικής πολιτικής και της ε, μπλε ανάπτυξης καθώς και 350.000 ευρώ για, την, για τους στόχους αυτούς κατά τη διάρκεια του παρόντος πρωτοκόλλου. Αναλαμβάνει επίσης ε, η χώρα αυτή να μπορέσει με αηφόρο τρόπο να εξασφαλίσει την ανάπτυξη των αλληλευτικών της πόρας. Η Επιτροπή Αλληλείας είναι υπεύθυνη επί και μας συνιστά να ψηφίσουμε το σχέδιο του Συμβουλίου σε σχέση με την ε, συμφωνία σύμπραξης που προβλέπεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κάπο Βέρτε. Από το, η διάρκεια του πρωτοκόλου αυτού του καινούργιου θα είναι εξαίτης 2019-2025. Ευχαριστώ. Θέλει κανένας από τους συναδέλφους και τους να λάβει τώρα το λόγο. Εάν όχι, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στην συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου. Έληξε λοιπόν η συνεδρίασή μας σήμερα, αλλά θα ήθελα να σας ε, καλέσω στις 3 ε, ε, Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες στο κοκτέιλ τέλους του έτους συνεδρίαση 3 Δεκεμβρίου στις 6 ώρα στις Βρυξέλλες. Κύριε Πρόεδρε, Δυστυχώς ε, ήμουν ε, κολλημένη στην κίνηση, είχαν ένα ατύχημα, κάτι φορτηγά εκεί στην, ε, στον αυτοκινητόδρομο. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ συγγνώμη για την αργοπορία, όμως θα ήθελα την Τετάρτη μετά, στην, μετά την ψηφοφορία να σας προσκαλέσω κι εγώ και να ευχαριστήσω όλους και όλες που έδειξαν τόσο μεγάλη υπομονή, που πολέμησαν, πάλεψαν μαζί μου και έδειξαν θάρρος. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσπάθειες που καταβάλλετε όλοι. Σα ευχαριστώ. Καλό σα βράδυ, εκτός από τους συντονιστέ οι οποίοι θα παραμείνουν στην αίθουσα. Non, excusez-moi,